Έξι προτάσει ψηφισμάτων έχω λάβει, έληξε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το τέλος τη συζήτηση. Η μερίσια διάταξη τώρα προβλέπει τη συζήτηση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέα. Μπαχρέιν, με συγχωρείτε. Ο Καρλ Σλέτερ έχει το λόγο. Βρισκόμαστε λοιπόν και πάλι εδώ, απέναντι σε μια χώρα όπου ένας λαός διεκδικεί τα δικαιώματά του, διεκδικεί την ελευθερία γνώμης, αυτό γίνεται ειρηνικά και μετά ακολουθεί η βίαιη καταστολή αυτή τη ειρηνική διαδηλώση. Αυτό το έχουμε δει συχνά το έργο. Σήμερα μιλάμε για το Μπαχρέιν. Όμως ε, το Μπαχρέιν έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχει πλέον ε, στο Μπαχρέιν ε, πίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν γίνει και οι σχετικές έρευνες. Εμείς όμως επιθυμούμε να υπάρχουν ανεξάρτητε αναλύσει. Επιθυμούμε να απελευθερωθούν όλοι οι ακτιβιστές. Δεν ξέρω βέβαια πόσε φορέ θα πρέπει να το δίκτυο επικίσουμε ακόμα αυτό από άλλες χώρες, όμως ε, στο ψήφισμα αναφέρονται και άλλα στοιχεία που μου αρέσουν πολύ. Παραδείγματος χάρη, εξαγωγές όπλων, οι εξαγωγές όπλων από τις ΗΠΑ προς τον Παχρέιν απαγορεύτηκαν. Είναι λοιπόν σημαντικό να καλέσουμε τώρα την Επιτροπή να τηρήσει αυτήν την απαγόρευση, αυτό το εμπάργκο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κερδίζουμε χρήματα με το να καταπιέζονται, να καταστέλλονται να καταπιέζονται μάλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καταστέλλονται οι ειρηνικέ διαδηλώσεις. Έχω κατά νου και τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες ε, στην περιοχή. Καλό λοιπόν την Επιτροπή να ελέγχει τις ε, εξαγωγές ε, όπλων. Επίσης πρέπει να προστατευτούν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαχρέν. Πρέπει να δρομολογηθεί στη χώρα αυτή η σχετική διαδικασία έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν η Αραβική Άνοιξη να μετατραπεί τελικά σε χειμώνα. Η κυρία Ντεκάιζερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αν νομίζουν ε, οι περισσότεροι δεν κάνουμε τίποτα την ε, πέμπτη το απόγευμα, δεν το πιστεύει το Μπαχρέιν γιατί πόσο γνωρίζω όλοι οι φίλοι που μετέβησαν στο Μπαχρέιν μας λέγανε ότι υπάρχει, επέρχεται μία αλλαγή, φυσάει ένας άνεμος αλλαγής, αλλά ε, θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς αποζητάμε με αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Όσοι διαδήλωναν ειρηνικά, οι ακτιβιστές, οι υπέρμαχοι της ειρήνης, γνώριζαν και γνωρίζουν ότι εδώ και ένα χρόνο μετά τα τραγικά γεγονότα επήλθαν αλλαγές και θα σας δώσω εντάχει δύο παραδείγματα. Η ανεξάρτητη επιτροπή που, ε, σύσταση, που, στην οποία, στη σύσταση της οποίας προέβη ο βασιλιάς μίλησε για βασανιστήρια, τα διαπίστωσε, για φυλακίσεις και ε, έγινε λόγος για παραδειγματική τιμωρία Επίσης υπάρχει μία τριμερής επιτροπή υπό τον ΔΟΕ με εκπροσώπους εργοδοσίας και εργαζομένων που έφτασε σε μία συμφωνία. Όλα αυτά είναι θετικά. Ίσως να μην αναφέρονται στο ψήφισμα, ας μην είμαστε όμως ιδιαίτερα αρνητικοί. Ας ε, πιστέψουμε σε αυτούς που θέλουν να επέλθει η δημοκρατία στο Μπαχρέιν, αλλά ας, είμαστε, ας επαγρυπνούμε κιόλας. Ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτά. Την, τον προηγούμενο μήνα ζητήσαμε τα ανθρώπινα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Και τότε υπήρχαν ενδείξει ε, ότι θα επενέβαινε η αστυνομία. Μετά από αυτό είχαμε την ε, επίμαχη άφηξη των ε, στρατευμάτων του GCC. Όμως ο Βασιλιά ξεκίνησε ένα διάλογο με τους διαμαρτυρόμενους και με το κόμμα της πλειοψηφίας του ΣΥΑ. Επίσης ε, πρότεινε και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ανησυχίες. Είπε ότι θα υπάρξει μια Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών στη χώρα ε, για να διασφαλιστεί η αποκατάσταση των ανθρωπιών δικαιωμάτων. Ε, και μάλιστα η ομάδα η δική μας καλεί τώρα τις αρχές του Μπαχρέιν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές αλλά να επιτρέψουν επίσης και την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη χώρα και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν οι έρευνες που γίνονται τώρα μπορούν να παρακολουθηθούν από εξωτερικούς συνεργάτες. Ε, όλα τα τεκτενόμενα θα ε, παρακολουθούνται από ανεξάρτητους ε, παρατηρητές. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή συζήτηση για την κατάσταση στο Μπαχρέιν, διότι αυτή η χώρα είναι από τις ε, ξεχασμένες της Αραβικής Άνοιξης. Η Αραβική Άνοιξη άρχισε εδώ και ένα χρόνο και μερικοί μίλησαν για μια επανάσταση που δεν θέλουμε να δούμε. Εμείς με τη σημερινή συζήτηση δείχνουμε ότι βλέπουμε την επανάσταση, ε, βλέπουμε την ε, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα καταδικάσουμε. Υπάρχει υπερβολική βία κατά των πολιτών και βεβαίως και άδικες δίκες. Καταδικάζουμε τους περιορισμούς των αρχών του Μπαχρέν κατά τον ΜΚΟ. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι στην κατάσταση και ζητούμε την παρακολούθηση της κατάστασης από την Ανεξάρτητη Επιστροπή. Η κυρία Βερσιά. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά, με συγχωρείτε, υπάρχουν ε, χώρες ε, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μελημάτων μας, όπως το Μπαχρέιν. Η επανάσταση κατεστάλλει βία και αυτό με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να καταδικαστεί και όχι μόνο να καταγγελθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία μερικών Πέρα από τις υποσχέσεις, οι καταστολές υπάρχουν. Και το είδαμε και στις 14 Φεβρουαρίου κατά τη μεγάλη διαδήλωση για την επέτειο του ενός έτους από την απαρχή της Επανάστασης. Όλοι σύρονται ε, στα δικαστήρια. Αυτό αφορά και τους ιατρούς που ε, περίθαλψαν τους διαδηλωτές. Πολλοί απολύθηκαν διότι συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες. Πολλοί σπουδαστές δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και η κυβέρνηση ζητά την αναβολή της επίσκεψης εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς ε, υπάρχει και ο πέμπτος στόλος των Αμερικανών που υποστηρίζει το Μπαχρέιν και άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι και οι ειδικέ δυνάμεις καταστολής, αστυνομικές δυνάμεις, είναι, διαδραματίζουν αρνητικό ρόλο. Αυτό μου θυμίζει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία θα πρέπει να, κάνουμε, να ασκήσουμε πίεση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για μένα αυτό το ψήφισμα πέρα από τις προσδοκίες μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εφόσον ε, είμαστε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να το δείξουμε ε, έμπρακτα. Η κυρία Σκάκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το φόρουμ στον Ταμπός φέτος χρηματοδοτήθηκε από τον Μπαχρέιν. Το Μπαχρέιν θέλει να εκλειφθεί σοβαρά από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον παγκόσμιο. Οι αρχές του Μπαχρέιν είναι αξιόπιστες μόνο όταν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελεία. Όταν η ελευθερία του λόγου περιορίζεται και το διαδίκτυο επίσης, η επιχειρηματική ανάπτυξη είναι αδύνατη. Όταν διαδηλωτέ ειρηνικοί έχουν να αντιμετωπίσουν βία και οι γιατροί έχουν να αντιμετωπίσουν πολιτικές δίκες, τα πράγματα δεν είναι ελκυστικά. Έχουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν στρατιωτικές δίκες και μπορεί να έχουμε και συμμετοχή του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Πρέπει οι απολυμμένοι να επαναπροσληφθούν και πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή όπλων προς τον Μπαχραήν. Το Μπαχραήν πρέπει να πάει στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να δείξει ότι πραγματικά σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Η, η απελευθέρωση του από του Χαγάτζα και από Άντι είναι πολύ σημαντική. Η απελευθέρωσή τους είναι πολύ σημαντική για την Ευρωβουλή. Ομάδα L, κυρία Μάκοβε. Έχουμε καταπίεση της των ειρηνικών διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν. Η κατάσταση χειροτερεύει παρά τις συστάσεις της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις. Συνεχίζεται η βία. Πεθάνανε πολλοί άνθρωποι λόγω του στρατιωτικού νόμου. Φτάσαμε στους 60 θανάτους που έχουν σχέση με γεγονότα το Δεκέμβριο. Οι αρχές του Μπαχρέν πρέπει να σταματήσουν να καταπιέζουν τις ε, διαδηλώσεις αυτές. Οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί επίσης δικάζονται απαράδεκτα στα στρατιωτικά δικαστήρια. Αυτές οι διώξεις πρέπει να σταματήσουν και οι οι αρχές που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες σωστής και δίκαιης δίκης πρέπει να είναι υπεύθυνοι για όσα πράττουν. Έχουμε καταστολή επίσης όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Υπάρχουν πάρα πολλοί αιστότοποι οι οποίοι είναι ε, μπλοκαρισμένοι στον Μπαχρέιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τιμήσει τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές. Ευχαριστώ κυρία Μακόβε. Η κυρία Γκέρνγκερ Ντεούντενμπεργκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι άνθρωποι του ο λαός μάλλον του Μπαχρέιν εμπνεύστηκε από τις ε, διαδηλώσεις στην Τινησία, στην Αίγυπτο, βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν διαδηλώσεις, επιδιώκουν μια συνταγματική μοναρχία να εγκαθιδρυθεί. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν βίων επιθέσεων 60 άνθρωποι πέθαναν εντωμεταξύ. Οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν να καταστέλνουν τον λαό τους, όλες τις ενέργειές τους, το διαδίκτυο επίσης και δεν επιτρέπουν το συνεταιρίζεστε. Ούτε καν την ελευθερία της μετακίνησης δεν επιτρέπουν των πολιτών. Ζητούμε λοιπόν οι πράξεις βίας αυτές να σταματήσουν άμεσα Ζητούμε οι θεμελιώδεις ελευθερίες να αποκατασταθούν και ένας επικοδομητικός διάλογος να αποκατασταθεί με την κοινωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ότζουλαν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μπαχρέιν έχει περάσει ήδη πολλές μεταβολές. Ε, Βεβαίω με τη θυσία πολλών αθώων πολιτών. Ε, αλλά έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση. Οι μεταρρυθμίσει όμω δεν μπορούν να υλοποιηθούν ε, όταν οι υπεύθυνοι για τα βασανιστήρια και τη δολοφονία πολιτών δεν δικαστούν. Ενθαρρύνω την κυβέρνηση του Μπαχραϊν να εγκαταλείψει τις καταγγελίες εναντίον ιατρών και διαδηλωτών να αποφυλακίσει τους φυλακισμένους και να ξεκινήσει ανεξάρτητες έρευνες για τις σοβαρές πράξεις βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Η κυβέρνηση του Μποχρέιν έχει διαπράξει πολλά σφάλματα και έχασε την αξιοπιστία, την αξιοπιστία της. Ελπίζω το δίδαγμα αυτό να τους αναποδώσει κάτι και να οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμίνσκι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχουν έθνη ή κράτη τα οποία δεν έχουν προορισμό να ζήσουν στη, με δημοκρατία. Η δημοκρατία παντού μπορεί να επιμερίσει. Γι' αυτό χαίρομαι για το κύμα μεταβολής που έφερε η, η Αραβική Άνοιξη. Ο αέρας αυτός φύσηξε και στον Παχραήν και πρέπει να σας πω ότι ο λαός του Παχραήν <clears throat> ήθελε και αυτός μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση ήθελε κάπως να υποχωρήσει. Υποσχέθηκε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Τα βήματα όμως, που, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Παχραήν δεν ήταν αρκετά. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Ε, όλα είναι πολύ ανησυχητικά ακόμη στο Μαχρέιν. Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι δεν έχουν πρόσβαση στο Μαχρέιν. Αυτό υποβαθμίζει την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία και δημοκρατία εάν άνθρωποι οι οποίοι διέπρεξαν δολοφιλνίες δεν δικάζονται. Ο κύριος Πάσκα τώρα για ένα λεπτό. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, πέρυσι στην Αραβική Άνοιξη υπήρξε αναταραχή και στον Μπαχρέν και σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Εκατοντάδες συνελήφθησαν. Ο βασιλιάς του Μπαχρέν συνέστησε Εθνική Επιτροπή και στην έκθεση διαπιστώνεται ότι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν ε, πέντε άνθρωποι. Ε, βία ασκήθηκε ε, έναντι των πολιτικών ακτιβιστών. Πολλοί άνθρωποι καταδικάστηκαν, όχι όμως με δίκαιη δίκη. Η Επιτροπή λοιπόν συνέστησε να υπάρξει μια Επιτροπή Έρευνας, να συσταθεί Επιτροπή Έρευνας, η οποία θα ερευνήσει τις υποθέσεις αυτές. Ε, πρέπει λοιπόν να ανανεωθεί η κοινωνική συνένεση, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες επικοδομητικού διαλόγου. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το γνωρίζει και ο Βασιλιάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς ε, η Αραβική Άνοιξη εντωμεταξύ έχει μετατραπεί σε αραβικό χειμώνα. Στον τύπο διαβάζουμε για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία, στη Λιβύη, ε, έναντι των κοπτών χριστιανών στην Αίγυπτο και τα γεγονότα στο Μπαχρέιν. Μόνο στο Μπαχρέιν από τότε που ε, ξέσπασαν οι σιητικές αντιδράσεις ε, έχουν δολοφονηθεί πάνω από 70 άτομα και το Σαββατοκύριακο η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα έναντι των ειρηνικών ε, διαδηλωτών και στρατεύματα της Σαουδικής Αραβίας στηρίζουν το καθεστώς του Μπαχρέιν με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν φροντίζουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις του καθεστώτος να είναι πιο ισχυρές από τις δυνάμεις της αλλαγής. Διαφυλάσσεται ο ζηλωτισμός με αυτά τα γεγονότα στο Μπαχρέιν ε, φθήνει και η ελπίδα να υπάρξουν δημοκρατικές διαδικασίες σε άλλα κράτη του κόλπου. Οι απαιτήσει του Μπαχρέιν για κοινωνική δικαιοσύνη, μεταρρυθμίσεις, ε, συνταγματική μοναρχία, ε, τα αιτήματα αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να κρίνουμε τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κύριος Κέλλη παρακαλώ. το Μπαχρέν δεν είναι η χειρότερη χώρα στον κόσμο, ούτε η πιο φτωχή, ε, ούτε πιο ε, καθυστερημένη. Παρόλα αυτά όμως τα θέματα που συζητάμε εδώ σήμερα είναι πολύ μεγάλη σημασία και ελπίζουμε ε, ως αποτέλεσμα το ψήφισμά μας θα σκίσει πίεση στις αρχές του Μπαχρέιν να προβεί στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η σύσταση αυτής της ανεξάρτητης επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη. Καλύτερα βέβαια θα ήταν να ληφθούν μέτρα με συγκεκριμένα αποτελέσματα κυρίως για τους ανθρώπους ε, που έχει διαπιστωθεί ότι διέπραξαν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξάλλου, ε, στον Μπαχρέν συνελήφθησαν άνθρωποι, ε, βασανίστηκαν θα πρέπει να αποκατασταθούν κυρίως εκείνοι που έχασαν τη δουλειά τους γιατί συμμετείχαν σε ειρηνικέ διαδηλώσεις. Και τέλος το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα πρέπει να πολλούνται όπλα στο Μπαχρέιν. Ευχαριστούμε. Ε, τώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye, η κυρία Εσάγια έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση ασφαλείας στο Μπαχρέιν παραμένει ε, κλειδονισμένη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία έντονη σύραξη και ε, δυστυχώς καταδιώκονται οι διαδηλωτές. Το Νοέμβριο ε, δημοσιεύτηκε μια έκθεση η οποία αναφέρθηκε στους συνεχείς βασανισμούς των διαδηλατών. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με την ε, Επιτροπή, την Ερευνητική Επιτροπή, πολλοί κρατούμενοι δυστυχώς βασανίζονται και ζητήθηκε να σταματήσουν αυτές οι δραστηριότητες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε απλώς ακροατές και θεατές αυτής της κατάστασης. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν, ότι έγιναν ορισμένα θετικά ε, βήματα αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ανεπάρκειες και δεν υπάρχει η κατάλληλη σπουδή για να διορθωθούν απαράδεκτες καταστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα στις Βρυξέλλες μία ομάδα γυναικών του Μπαχρέιν που μου είπαν ότι δυστυχώς χειραγωγήθηκαν. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν δρά η κυβέρνηση του Μπαχρέν. Γιατί ο ειδικό εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανισμών δεν δρά. Γιατί το Μπαχρέιν δεν ζήτησε οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών να επισκεφθούν τη χώρα. Μέσω της ΥΠΑ της εκπροσώπου θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Μπαχρέιν να προβεί στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και να τηρήσει την ε, κοινή θέση ως προς την ε, εξαγωγή όπλων έτσι ώστε να μην είμαστε και εμείς συνένοχοι αυτής της κατάστασης τη στιγμή που εξάγουμε όπλα. Η κυρία Νικολάη Νομίζω ότι το Μπαχρέιν μας δείχνει ότι προτρέξαμε ως διεθνής κοινότητα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Πέρσι μιλήσαμε για θετικές ενέργειες και είπαμε, ελέγχθη ότι ότι δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνέχεια ο βασιλιάς διόρισε μία άλλη επιτροπή για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτό, αυτή η έκθεση θα υποβληθεί στις 20 Μαρτίου και θα δούμε τι θα γίνει. Όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις πιέσεις μας για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση ψηφίσματος και νομίζω ότι μόνο με πιέσεις μπορούμε να επιτύχουμε κάτι το θετικό. Η κυρία Κορόλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τον Οκτώβριο είδαμε πώς είχε η κατάσταση στον Μπαχρέιν, την εξέλιξή της. Διαβάσαμε πολλά για, για αυτούς που εργάζονται σε νοσοκομεία να συλλαμβάνονται παραδείγματο χάρη επειδή είχαν φροντίσει τραυματισμένους από τις διαδηλώσεις. Αυτές είναι ειρηνικέ διαδηλώσεις, δεν είναι βίες. Λοιπόν, πρέπει να επικεντρωθούμε στα σοβαρά και πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τον αποκλεισμό των πολιτών από τις διαδηλώσεις. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις αναμφισβήτητα. Χρειάζεται και σωστή αντιμετώπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων αυτών που προσπαθούν να φέρουν κάποια αλλαγή. Ο Σουλτάνος του Μπαχρέιν και οι αρχές μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν την πρόθεση να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους. Ο κύριος Ρέπο, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ο λαός του Μπαχρέιν ζητάει δημοκρατική μεταρρύθμιση και το σεβασμό των θεμελιωδιών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης επίσης. Αυτές δεν είναι υπερβολικές απαιτήσει ούτε και απειλή κατά της κυβέρνησης του Μπαχρέιν. Αντί να ανταποκριθεί λοιπόν η κυβέρνηση εκεί, η ε, ασφάλεια συνέχισε να επιτίθεται κατά των διαδηλωτών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιούνται η μέσα κατά άμαχων και άοπλων διαδηλωτών. Είναι δικαίωμά τους να διαδηλώνουν, καθώς και η κοινωνία των πολιτών. Η κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει την δραστηριοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών οι διαδηλώσεις επιδιώκουν περισσότερη δημοκρατία, δραστηρι... ενέργειες και δραστηριότητες ώστε να δημιουργηθούν θέσει εργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο τελείωσε. Κυρία Πρόεδρε, εγώ τον Μπαχρέν το ξέρω εδώ και 30 χρόνια και θέλω να σας πω ότι η χώρα αυτή ήταν σε πολύ καλό δρόμο και μπορεί να επανέλθει στο σωστό δρόμο και αυτό παρά το ότι ε, είναι εκτεθειμένο απέναντι στο Ιράν. Βεβαίως ε, και υπάρχουν ε, επιθέσεις της εξουσίας ε, και των ε, Σαουδαράβων ε, που βρίσκονται πίσω από τον Μπακρέιν που θα ήθελαν πολύ ευχάριστα να το προσαρτήσουν. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια συστηματική σιητική αναταραχή που εξωθείται από το Ιράν και από τους ακραίους ηγέτες του Ιράν. Και τα δύο είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και το δικό μας το καθήκον δεν είναι να είμαστε μονομερείς αλλά να μεσολαβούμε έτσι ώστε να υπάρχει στη χώρα αυτή μια εύρυθμα λειτουργούσα συνταγματική ε, μοναρχία, μια ισορροπία ανάμεσα σε Σιήτες και Σουνίτες, γιατί αλλιώς θα υπάρξει αναπόφευκτη αιματοχυσία. Η αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη δυστυχώς ε, στις περισσότερες χώρες τώρα τίνει να εξελιχθεί σε ε, ακραίες, σε καταστάσεις. Και αυτό νομίζω το εκμεταλλεύονται και οι ακραίοι στο Μπαχρέιν. Τελευταία μιλήτρια, η κυρία Τάιν. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω το ότι το κοινοβούλιο αυτό ασχολείται με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν. Ε, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν έχει δημοσιεύσει έναν κατάλογο α, δολοφονημένων και ο κατάλογος αυτός είναι πολύ πιο μακρύς, 66 αναφέρονται οι νεκροί. Η συζήτηση είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό κρατών, ε, κράτη τα οποία σιωπούν μπροστά σε αυτά που διαδραματίζονται στο Μπαχρέιν και θα έπρεπε ανταυτού να υψώσουν τη φωνή τους. Αν δει κανεί ε, τις αντιδράσεις ε, των κρατών μελών τότε που είχαμε τους πρώτους νεκρούς στη Συρία εκεί η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική. Ελπίζω λοιπόν τουλάχιστον σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εφαρμόζονται παντού τα ίδια μέτρα και σταθμά ανεξάρτητα από τη χώρα. Όχι δηλαδή επειδή στο Μπαχρέιν έχουμε αμερικανική βάση στόλου και όχι ρωσική. Όχι επειδή στέλνονται και αμερικανικά και όχι ρωσικά όπλα και όχι επειδή έχουμε καλύτερες εμπορικές σχέσεις με τον Μπαχρέιν από ότι με τη Συρία να κρίνουμε τα πράγματα διαφορετικά πρέπει παντού να κρίνουμε με τέτοια μέτρα και σταθμά όταν πρόκειται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος. Α, με συγχωρείτε κυρία Επίτροπε, σα ξέχασα, σας ξέχασα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει μεγάλη προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν. Ιδιαίτερα καθώς μια ε, έγινε μια έρευνα από τον περασμένο Φεβρουάριο σε αυτή τη χώρα. Αυθαίρετες συλλήψεις, κακή μεταχείριση, ακόμη και βασανιστήρια συλληφθέντων διαπιστώσαμε. Δίκες χωρίς εγγύησης και χωρι... Ε, περιορισμός των θεμελιών δών ελευθεριών. Πρέπει να βελτιωθούν λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία συμφιλίωσης εθνικής. Είναι ανησυχητική η κατάσταση και η απόκριση πάντα υπήρξε ίδια. Η κάθε Άστον, το αντιπρόσωπος, εξέδωσε έξι δηλώσεις την ε, τον περασμένο χρόνο για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Έθεσε πολλές φορές αυτό το ζήτημα στον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν και συνάντησε και τον ίδιο τον Βασιλιά τον Απρίλιο η Επιτροπή, το Συμβούλιο με συγχωρείτε εξωτερικών υποθέσεων επανέλαβε τα ίδια μηνύματα το Μάρτιο και το Μάιο και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ριάντ που είναι διαπιστευμένη και στο Μπαχρέιν έχει διάλογο με τις αρχές η Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρεται για την απόφαση του Βασιλιά τον Ιούνιο του 2011 να θέσει να δημιουργήσει ανεξάρτητη επιτροπή εξεταστική ε, για τις διαδηλώσεις, για την αναταραχή. Ε, οι συστάσεις αυτής της Επιτροπής εφαρμόζονται τώρα από την κυβέρνηση. Δημοσιεύθηκε η έκθεση τον Νοέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε προθυμία να υποστηρίξει συγκεκριμένα την κυβέρνηση του Μπαχρέιν ε, για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτές τις προσδοκίες. είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις πλήρως και είναι εξίσου σημαντικό να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των αρχών και της αντιπολίτευσης. Οι ομάδες της αντιπολίτευσης πρέπει και αυτές να παίξουν το δικό τους ρόλο για να το καταστήσουν εφικτό. Διότι αν δεν υπάρξει διάλογος δεν θα υπάρξει και διαρκής εθνική συμφιλίωση. Τέλος, ελπίζουμε ότι οι ποινές που έχουν επιβληθεί από τα δικαστήρια εθνικής ασφάλειας όπως αποκαλούνται σε ομάδα 20 γιατρών και πολλών υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ανακληθούν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν από νέα δίκη ε, ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων με όλες τις απαραίτητες εγγυήσει βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Σας ευχαριστώ. Όπως σας έλεγα, κάπως πρόωρα. Α, κυρία Γκόμες, συγγνώμη. Διαδικαστικό. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι αναφέρεται στα μέσα ενημέρωση ότι η Αιθιοπία επιτέθηκε στην Ερυθρέα, πολλοί ε, δολοφονήθηκαν και δύο, ε, είχαμε και δύο απαγωγές. Ξέρετε αυτές οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε ματηρό πόλεμο τη δεκαετία του 90. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γιατί όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την Αιθιοπία αλλά και ε, δεν έχει επιβάλει το σεβασμό των συνόρων, κάτι που αποφασίστηκε πριν από κάποια χρόνια. Αυτό είναι υπέρ της Αιτιοπίας. Θέλω λοιπόν μέσω ημών ε, να καλέσετε την κυρία Άστον να έρθει την άλλη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει ε, σε αυτές τις ε, δύο χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πόσελτ. Κυρία Πρόεδρε, μόλις και εγώ ε, ενημερώθηκα ότι ε, το, η επόμενη Ολομέλεια θα ξεκινήσει την Τρίτη λόγω του Ορθόδοξου Πάσχα και θα πάμε μέχρι την Παρασκευή. Η διάσκεψη των Πρόεδρων αποφάσισε να ε, αφαιρέσει τα κατεπήγοντα από την εμμυρίσια διάταξη. Αυτό δεν είναι σωστό. Στις τέσσερις εβδομάδες μέχρι την Ολομέλεια του Απριλίου θα προκύψουν πολλά και επίγοντα θέματα. Εγώ λοιπόν διαμαρτύρομαι. Διαμαρτύρομαι γιατί λαμβάνονται αποφάσεις που παραβιάζουν τους κανόνες μας και παρακαλώ τους αδέλφους από άλλες πολιτικές ομάδες να μιλήσουν και αυτοί με τους επικεφαλής για να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση μέχρι τον Απρίλιο. Ε, λαμβάνω υπόψη τα σχόλια σας. Ε, βεβαίως η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφανθεί, θα διαβάσουμε το έτοιμά σας στη διάσκεψη. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση, λίγη η συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος. Η συζήτηση έχει λήξει και περνάμε στην